για την καταπολέμηση της απάτης στην Ολομέλεια γιατί ίσως ε, θεωρείτε ότι το ένα θέμα σχετίζεται άμεσα με το άλλο. Ναι, θα συμπεριληφθεί η ομιλία σας. Θα συμπεριληφθεί σε αυτό το σημείο της σημερινής διάδευσης και όχι στο προηγούμενο. Δεν εργαστήκατε εις την κυρία Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ, λέγει η κυρία Μπασέσκου. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 6 από τις 9 μέχρι τη 1. Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη στο ίντρανετ. Λύεται η συνεδρίαση σας. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Χαίρετε.